Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα για τις επιπλέον πληροφορίες. Περνάμε τώρα στην ανακοίνωση της παρέτησης του Παύλο Ιγλέσιας και του Φερνάντο Μάουρα Μπαραντιαράν. Σύμφωνα με τον κανόνα, με τον άρθρο του κανονισμού, ε, οι θέσεις θα κηρυχθούν χειρεύουσες από τις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Νοεμβρίου διαδοχικά